Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt Ruhe zu geben. Please sit down and be quiet. Κυρίες και κύριοι, σας καλώ να καθίσετε όλοι και να κάνετε ησυχία. Σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία, ειδικότερα εκεί στις θέσεις των βοηθών ησυχία. Äh, θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω εγκάρδια. Κύριε Πρωθυπουργέ. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω εγκάρδια ε, εδώ στις Βρυξέλλες κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή σας, εδώ λοιπόν στο πλαίσιο της δικής μας ε, Επιτροπής ε, σε συνεργασία με την άλλη Κοινοβουλευτική Επιτροπή σας έχουμε καλέσει λοιπόν εδώ και θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στους πρόεδρους αυτών των δύο επιτροπών μετά από μένα για να απευθυνθούν σε εσά. Νομίζω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί αυτή την περίοδο της εξελίξης στη χώρα σας ε, με μεγάλο ενδιαφέρον και ε, προσπαθεί βέβαια από την πλευρά του να ενισχύσει και τη ε, δημοκρατική εξέλιξη. Μιλάμε για μία από τις χώρες με την οποία έχουμε πολύ εντατική συνεργασία και συνάδελφος έχει αναλάβει και μια στενή συνεργασία στο πλαίσιο των αποστολών για την υποστήριξη της δημοκρατίας, τα Democracy Support Missions και νομίζω πως θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι πραγματικά οι εξέλιξη ε, στην Τινησία είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρε σε σύγκριση με άλλε χώρε τη ίδια ε, περιοχή. και θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε από εσά το πώ πηγαίνουν τα πράγματα, πώς βλέπετε εσεί τι ε, προοπτικές. Αλλά βέβαια το να υπάρχει μια τέτοια θετική εξέλιξη στην Τινησία είναι και προ το δικό μα συμφέρον. Όντως ώστε δηλαδή οι σχέσει μα. Ε, να γίνουν ε, σχέσεις οι οποίες μας ενώνουν, όχι μας χωρίζουν και εδώ αναφέρομαι βέβαια στις ε, πολιτικές γειτονίας. Η σχετική πολιτική γειτονία θα πρέπει νομίζω να αναδιαμορφωθεί ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στα εκείνα μας συμφέροντα και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να κινηθούμε. Επίσης μας ενδιαφέρουν συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα ε, Πρόεδρο, από ό,τι γνωρίζουμε, έπρεπε στη σύναψη μια συμφωνία με τι ε, ε, ΗΠΑ ω ε, μείζον ε, σύμμαχος ε, του ΝΑΤΟ. Θα θέλαμε να ακούσουμε και το τι ακριβώ εμπεριέχεται σε αυτήν την συνεργασία και το πώ μπορούμε περαιτέρω να αναπτύξουμε και τη συνεργασία σα με την Eurojust και με την Europol. Επίσης θα θέλαμε να ακούσουμε βέβαια και ποια είναι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα σας γιατί προφανώς είναι σημαντικό να υπάρχει μια ε, πολύ καλή οικονομική και κοινωνική κατάσταση, ούτως ώστε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και ταυτόχρονα ε, βούληση για ε, επενδύσεις, τις οποίες βέβαια χρειάζεται ιδιαίτερα η χώρα σας. Και προκειμένου να επιτευχθεί και η υπεραξία τέτοιων επενδύσεων. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να ενισχυθεί η δημοκρατική διαδικασία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που έχετε προσέλθει σήμερα εδώ Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Βερσιάνου για να απευθυνθεί και εκείνη. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σίδ. Ευχαριστώ, κύριε Σαριφάτ, που ήρθατε σήμερα να επισκεφτείτε το κοινοβούλιο μας και να ανταλλάξουμε μαζί πληροφορίες όσον αφορά τις πιο πρόσφατες ε, καταστάσεις στη χώρα σας συμμετείχα και εγώ στην αντιπροσωπή για την παρατήρηση των εκλογών και εντυπωσιάστηκα και συγκινήθηκα μπορώ να πω από τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην Τινησία. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο ατού η κοινωνία των πολιτών. Το κοινοβούλιο μας έχει δεσμευτεί να στηρίξει το δικό σας κοινοβούλιο ένα από τα συμπεράσματα στην ε, έκθεση της αποστολής παρατήρησης των εκλογών, ένα από τα συμπεράσματά μας ήταν να συνεργαστούμε με τους βουλευτές της Τινησίας και κυρίως με τους πιο νέους και τις γυναίκες βουλευτές και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες στιγμές για να ανταλλάσσουμε απόψεις, πληροφορίες ίσως, να έχουμε ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών. Προτείνω λοιπόν πραγματικά αυτό να κάνουμε να λάβουμε υπόψη μας τη σύσταση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που ήρθατε και σας συγχαίρω για το έργο σας. Η Τινησία αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Μεσόγειο και έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να σας στηρίξουμε. Και πάλι συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ. Κύριε Μπρόκ, τελείωσα. Das Wort hat Κύριε Φωτίγα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ε, διερμηνείς αν είναι δυνατόν να μιλήσω στη γλώσσα μου. Ε, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξή. Νομίζω πως έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Έχουμε πάρα πολλά κοινά με τον Πρωθυπουργό της Τινησίας. Ο κοινός πολλαπλασιαστής ε, έγκυται στην προσπάθειά μας προς τους δημοκρατικούς θεσμούς και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Μεσόγειος πρωτίστως που είναι ο βασικός μας σύνδεσμος και η γέφυρα που μας συνδέει γενικότερα. Έχω μία ερώτηση να σας υποβάλω. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να καταβάλει προσπάθεια κατά των διακινητών ανθρώπων και έχουμε προβεί στη σύσταση θαλάσσιων επιχειρήσεων. Ποια είναι η γνώμη σας για τις θαλάσσιες αυτές επιχειρήσεις και ποιες είναι οι επιλογές που διαθέτει η Τινησία του θέματος. Honorable député, mesdames et messieurs. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ και απευθύνομαι στο σώμα σας και θέλω επί τη ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις όσον αφορά τις εξελίξεις στην Τινησία και τις προοπτικές της χώρας προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου επίσης να χαιρετήσω εδώ το ρόλο και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως χώρος δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλω να επιθεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να ευχαριστήσω για τη στήριξή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στήριξη που μας προσφέρει από το 2011 μετά από την δημοκρατική εμπειρία στην Τινησία. Με οικουμενικές αξίες, την ελευθερία, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές και όλους τους υπεύθυνους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκονται εδώ παρόντες για την δέσμευσή τους να στηρίξουν την Τινησία. Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, μετά από την τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ στις Βρυξέλλες το 2011, θα θυμόσαστε και το ξέρετε ότι έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στην Τινησία που μας επέτρεψαν να εγκαινιάσουμε μια νέα περίοδο στην ιστορία της χώρας μας. Να γυρίσουμε μια νέα σελίδα. Βέβαια, στις 27 Ιανουαρίου του 2014 είχαμε το νέο σύνταγμα. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε η δεύτερη δημοκρατία στην Τινησία, κάτι που σημαίνει ότι ο τη της αν ανεπιστρεπτή είναι υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Το Σύνταγμα αφιερώνει ένα κομμάτι στην, στο λεκό χαρακτήρα της χώρας υπέρ του κράτους δικαίου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης αναφέρονται και οι προδιαγραφές οι δημοκρατικές. Και πρόκειται για τις βάσεις μια συμμετοχικής δημοκρατίας χωρίς αποκλισμούς τόσο σε εθνικό όσο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τον Οκτώβριο του 2014 είχαμε εκλογέ κοινοβουλευτικέ και τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο εκλογές που μου δίνουν την ευκαιρία να εκφράσω και πάλι την εκτίμησή μου για την στήριξή σας, τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της αποστολής σας παρατήρησης των εκλογών αυτών. Οι εκλογές ε, αυτές, ελεύθερες, με διαφάνεια, και σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές, όπως χαρακτηρίστηκαν από τους παρατηρητές, σε όλα τα επίπεδα, μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε την διαδικασία μετάβασης, μεταπολίτευσης και να έχουμε θεσμούς ε, σήμερα που βασίζονται στο κράτος δικαίου. Όπως γνωρίζετε, οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν κάτι εύκολο για μας. Παρ' όλα αυτά, ο λαός της Τινησίας έδειξε ότι προτιμάει το διάλογο και την συνένεση. Και έτσι προχώρησε στη δημοκρατική διαδικασία. Είναι μια εμπειρία χωρίς προηγούμενο στο περιφερειακό επίπεδο, η οποία φέρει καρπούς για όλους τους τινήσιους, σύμφωνα με τις αξίες της ανοχής, της μετριοπάθειας, και μη αποδοχή του εξτρεμισμού και της βίας. Κυρίες και κύριοι, οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα μαρτυρούν, είναι αλήθεια, μεγάλες πολιτικές αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα και μαρτυρούν επίσης και το δυναμισμό των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα συνεχιζόμενο έργο, σε καθημερινή βάση, που απαιτεί τη συνεργασία όλων των δυνάμεων της χώρας. Σήμερα Μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκεται η χώρα, η πολιτική αυτή διαδικασία πρέπει να προστατευτεί και το δημοκρατικό οικοδόμημα να ενισχυθεί. Πρώτα απ' όλα έχουμε την πρόκληση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης την πρόκληση αυτή πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Η, οικονομική ανάπτυξη περνάει από ξένες επενδύσεις, από ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, από τη δημιουργία απασχόλησης, κυρίως για τους νέους διπλωματούχους με πτυχίο πανεπιστημίου και την κατάργηση των ανισοτήτων. Θέλουμε επίσης κοινωνική ειρήνη. Όλα αυτά αποτελούν βάση για την οικονομική μας ανάκαμψη. Η ασφάλεια έπειτα. Επίσης αποτελεί μεγάλη πρόκληση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι στο κέντρο της δράσης μας δεδομένης ε, της κατάστασης στην περιοχή. Η Τινησία που είναι θύμα δηλών τρομοκρατικών ενεργειών είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της για να ξεριζώσει την απειλή αυτή. Όμως είναι βέβαιο ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού γράφεται σε μια γενικότερη προσέγγιση. Χρειάζεται μια συνοχή που ξεπερνάει τα όρια της ασφάλειας και περνά και μέσα από την κοινωνική διάσταση, την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την προληπτική. Πρέπει επίσης να βασιστούμε σε μια συνολική προσπάθεια και τη δέσμευση όλων χωρών και εταίρων. Η κατάσταση στη Λιβύη, για παράδειγμα, πρέπει να τακτοποιηθεί για να υπάρξει σταθερότητα τόσο στην ίδια τη Λιβύη αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Γι' αυτό και πρέπει σήμερα να συνδυάσουμε όλες τις προσπάθειες που μπορούμε για να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να πετύχει ο διάλογος στη Λιβύη και να μπορέσει η χώρα να καταλήξει σε μια ειρηνική λύση της ε, κρίσης που τη μαστίζει σήμερα. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, εμβάθυνση της εταιρική σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που αποτελεί ιστορική σημασία σε επιλογή και στρατηγική για την Τινησία. Έτσι η Τινησία τα τελευταία χρόνια έχει νιώσει την βοήθεια αυτή από τη δικιά σας την πλευρά με επαφές σε όλα τα επίπεδα, με τις επισκέψεις που κάνατε. Δείχνει επίσης τις διάφορες δράσεις συνεργασίας που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης και οι θεματικές συνεδριάσεις που έγιναν, που αποτελούν πολύ καλές ευκαιρίες για να συζητούμε μαζί με επικοδομητικό πνεύμα συγκεκριμένα μέσα για να ενισχύσουμε τις ανταλλαγές μας η προτιμησιακή αυτή η εταιρική σχέση το 2014. Εγγράφει έτσι τις σχέσεις μας σε ένα όραμα στρατηγικής σημασίας, με διάρκεια υπέρ των αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τις οποίες συμφωνούμε απόλυτα. Επίσης ανοίγει νέες προοπτικές για την ενίσχυση της συνεργασίας και σε καινοτόμους τομείς. Έτσι λοιπόν θέλω εδώ σαν παράδειγμα να δώσω διάφορα παραδείγματα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της προτιμησιακής αυτής εταιρικής σχέσης. Στα τέλη του Απριλίου του 2015, επί τη ευκαιρία του Επιτρόπου Χάνα στην ε, την υπογράψαμε πέντε οικονομικές συμφωνίες που καλύπτουν διάφορους τομείς και είναι κάτι το οποίο μαρτυρεί για άλλη μια φορά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τινησία για τις μεταρρυθμίσεις της. Επίσης, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το νέο πρόγραμμα στήριξης για την εσωτερική ασφάλεια της Τινησίας, κάτι το οποίο αποτελεί, δεδομένης της σημερινής κατάστασης, ένα σημαντικό πρόγραμμα, ένα εμβληματικό πρόγραμμα. Η συνεργασία μας διευρύνεται επίσης και σε άλλους τομείς ασφάλεια στην Τινησία. Για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο, η μεγάλη αυτή πρόκληση, η Τινησία χρειάζεται τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ μιας μεγαλύτερης εμπλοκής των ευρωπαϊκών θεσμών και τεχνικά και οικονομικά, προκειμένου να αναπτυχθεί η χώρα. Χρειάζεται μια δέσμευση από την πλευρά σας που να συνάδει με τις μεγάλες φιλοδοξίες που συμπεριλαμβάνονται στην εταιρική μας σχέση και να είναι και στο ύψος της μοναδικής δημοκρατικής εμπειρίας της Τινησίας. Εξίσου σημαντικό είναι εδώ να υπογραμμίσουμε και την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γυτνίασης. Η αναθεώρηση αυτή πρέπει να εγγράφεται στα πλαίσια μιας γενικής προσέγγισης των σημερινών μας και μελλοντικών μας σχέσεων. Μια προσέγγιση που πρέπει να πηγαίνει προς μια κοινή άποψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να ληφθούν υπόψη διατερότητες μας. Ένα ένας κοινός στόχος η Μεσόγειος να γίνει χώρο συνοχής, αλληλεγγύης και ειρήνης. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου τέλος να επαναλάβω την εκτίμησή μου για την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Τινησία, προς τη νέα αυτή δημοκρατία, η οποία αξίζει για την ε, περίοδο που έρχεται την προσοχή σας και τη φιλία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριος Πρίδιος, πρώτος ο μιλητής. Σας καλωσορίζω και εγώ κύριε Πρωθυπουργέ εξ ονόματος του ΕΛΚ. Θα ήθελα να σας πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί μπορούμε να προβούμε σε ανταλλαγές απόψεων μαζί σας σήμερα στα πλαίσια μιας γενικότερης σκέψης για την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας. Και ήδη έγιναν ανταλλαγές απόψεων για την ανάγκη μεγαλύτερες, μεγαλύτερης ευελιξίας για την πολιτική γειτονίας για να κατανοήσουμε το δρόμο που πρέπει να διανύσει κανείς από πλευράς βορρά και νότου ο εισηγητής μας θα επανέλθει επί του θέματος. Θα ήθελα να σας πω επίσης ε, ότι χαιρόμαστε γιατί είδαμε και τις πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα σημαίνουσες στη χώρα σας, ιδιαίτερα την πολιτική διαδοχή αυτή, η εναλλαγή που εγκαθιδρεί τη δημοκρατία και συγχαίρω τον λαό της Τινησίας γιατί είχε αυτή την δυνατότητα και τη χρησιμοποίησε. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για την απαρχή αυτής της διαδικασίας των θυμάτων της δικτατορίας, ε, των βασανιστήριων, της κατάχρησης, των καταχρήσεων, δηλαδή αυτής της ε, μεταβατικής ε, δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ όλοι οι ομιλητές να τηρήσουν το χρόνο των δύο λεπτών. Ε, και επιτρέψτε μου τώρα να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Αλλιώ δεν θα προλάβουν να μιλήσουν όλοι. Ο κύριο Παγνού, ω επόμενο ομιλητή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχήν να σας καλωσορίσω και εγώ σε αυτή την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ευγενικά σας λόγια και για όσα Λέτε εδώ και τέσσερα χρόνια από το 2011 αυτή η δημοκρατική βιτρίνα ε, τιμά και εμάς και μια χώρα όπως η Ισία. Αυτά τα χρόνια ζήσαμε αυτή την δημοκρατική μετάβαση και δημοκρατική ζωή στη συνέχεια η οποία έχει παγιωθεί πλέον σήμερα με τις ε, δράσεις σας, με τη δράση σας γενικότερα, τον μεν και τον δε, στη μεγάλη αυτή χώρα που λέγεται την Ισία. Όπως είπατε, πέρα από αυτή τη δημοκρατική εικόνα προς τα έξω, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, εταιρική μας σχέση. Τον Απρίλιο του 2005 υπογράψαμε πέντε συμβάσεις και αυτό που έχει σημασία είναι και η ασφάλεια με τη γείτονα χώρα, τη Λιβύη και τη δημοκρατική διαδικασία που έχει ξεκινήσει και εκεί, αλλά και στην Τινήσια. Δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε ότι το χάος στη Λιβύη διεισδύει και στην Τινησία και δημιουργεί παράδοξες καταστάσεις. Μάθαμε ότι στις 18 Μαΐου 512 την ίση συνελήφθησαν στη Λιβύη και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η δική σας κυβέρνηση και η κυβέρνηση της ε, Τρίπολης βρίσκονται σε μια κατάσταση διελκυστίνδας μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, περιφερειακής διένεξης Πώς ε, μπορείτε να αποφύγετε τη διένεξη με την κυβέρνηση του Τομπρούκ που αναγνώρισε η διεθνής κοινότητα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μία ομοιογένεια και στα, στα δυτικά της χώρας, με, στα πλαίσια και του Ζιντάν, προς δυσμάς της Λιβύης. Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Σας παρακαλώ να παραμένετε στα δύο λεπτά. Να είστε ε, σωστοί απέναντι στους συναδέλφους. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά, όχι δύο λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, όπως στη δική σας περίπτωση. Ο κύριος Τάνοκ θα μας το αποδείξει αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ να σας ε, ευχαριστήσω εξ ονόματος του ECR. Εγώ πάντα ήμουν φίλος της ε, Τινησίας και θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη μεγάλη σας επιτυχία κατά την Αραβική Άνοιξη και την νίκη του κόμματός σας ε, πέρσι τον Οκτώβριο περνώντας σε ένα κοσμικό καθεστώς. Τα καταφέρατε με τις εκλογές και αυτό είναι εξαιρετικό. Οι ερωτήσεις μου έχουν ως εξής. Ως προς ε, την κατάσταση της Λιβύης ε, βρέθηκα με τον πρέσβη μας ε, στη Λιβύη, ο οποίος ζει στην την Ισία για την κατάσταση στην Τρίπολη. Είναι πολύ επικίνδυνη. Στην Ιταλία μάθαμε ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος ε, της ε, τρομοκρατικής ενέργειας στο Μουσείο της Τινησίας, ο οποίος έφτασε σε, με ένα πλοίο από αυτά που μετέφερε τους, ε, μετέφεραν τους μετανάστες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα του να διεισδύσουν τρομοκρατικά στοιχεία στην Ευρώπη προβάλλοντας ε, μάλλον μέσα στα πλαίσια των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, πώς ε, μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα των διακινητών μέσα στα πλαίσια του ψηφίσματος της απόφασης 7 των Ηνωμένων Εθνών και πώς ε, μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους διακινητές μέσα στα πλαίσια των χωρικών σας υδάτων. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ένα ε, καθεστώς τύπου, μια επιχείρηση τύπου Ατλάντα στη Σομαλία. Ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του Μπέναλι πώς ε, μπορείτε να ανακτήσετε αυτά τα κτήματα από χώρες μεταξύ των ε, οποίων και από, την, από το Ηνωμένο Βασιλείο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά, Φλαμανδικά, αν μου επιτρέπετε. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας καλωσορίσω που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε ένα τέτοιο Πρωθυπουργό και να τον ακούμε να μιλάει για μια χώρα που παίζει σημαντικό ρόλο. Η Τινησία είναι και εμπορικό εταίρο και γείτονα τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε πολύ κοντά. Η χώρα σα επίση μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή, μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό παράδειγμα για του γειτονέ σα νοτιότερα μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για τη σταθερότητα στην περιοχή που τόσο πολύ τη χρειάζεται. Τα αποτελέσματα επίσης τα εκλογικά το 2014 είναι σημαντικά στη χώρα σας. Νέο σύνταγμα, δημοκρατικές αξίες, στη χώρα σας. Πολύ σημαντικό. Οι εκλογές ε, επίσης έλαβαν χώρα χωρίς προβλήματα, με διαφάνεια. Υπάρχει ένα κράτος δικαίου, δικαιοσύνη που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο βάσει των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών. Μόνο θετικά σχόλια έχει κανείς να κάνει. Αλλά βέβαια υπάρχουν και ερωτήσεις για τη χώρα σας. Εξάλλου γι' αυτό σας φωνάξαμε να έρθετε εδώ και σας καλέσαμε. Υπάρχουν ε, ακόμα δημοσιογράφοι και αγωνιστές οι οποίοι κινδυνεύουν με φυλάκιση επειδή ε, ασκούν την ελευθερία έκφρασης, αυτό το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, θέλω να μάθω την απόψή σας. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις αυτές και τι γίνεται με την ελευθερία έκφραση στη χώρα σας. Μια που υπάρχουν επικριτικές φωνές από αυτού. Δεύτερον, είμαστε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο όπου όπως ξέρετε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι τις τεράστιες μεταναστευτικές ε, ροές. Τι γίνεται λοιπόν με τα πλοία εκείνα τα οποία φορτώνουν τους μετανάστες προς τις χώρες και πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Είμαι φίλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Τινησιακού λαού. Έχω συμμετάσχει σε όλες τις αποστολές ε, παρατήρησης των εκλογών από το 2011. Έχω παρακολουθήσει τις δυσκολίες αλλά και την μεγάλη δυνατότητα που έχετε για αλλαγές. Η κυρία Βαλενθιάνο εξάλλου το είπε ότι η κοινωνία των πολιτών σας είναι ένα τεράστιο ατού για να σας συνοδεύσει στις αλλαγές ε, αυτές κάθε φορά που χρειάζεται. Η Τινησία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σε περίπλοκη θέση, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν αποτελεί σημείο αναφορά παράδειγμα ή δεν ξέρω τι, πολλά ακούσαμε αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει την Τινησία στην κατάσταση ακριβώς την ιδιαίτερη αυτή που βρίσκεται και πρέπει να το κάνει με φυή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τι διακυδεύεται πολιτικά σε ολόκληρη την περιοχή. Σήμερα έχετε σταθερούς θεσμούς, αλλά παραμένουν πολλά να γίνουν οικονομικά, κοινωνικά, πρώτα απ' όλα, γιατί οι λόγοι που οδήγησαν στην ε, στις αλλαγές το 2011 στην Τινησία παραμένουν. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, υπήρξαν 100 κοινωνικές ε, συγκρούσεις τον τελευταίο καιρό. Η Κάφσκα, Ρεβέγεφ, εκεί όπου άρχισαν τα προβλήματα, παραμένουν να έχουν τα ίδια προβλήματα. Πολλές είναι οι προσδοκίες, ε, οι ελπίδες της νεολαίας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ακόμα μια τεράστια προσπάθεια. Διάβασα διάφορα, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η προτεραιότητα θα είναι ο κοινωνικό διάλογο. Κάτι πολύ βασικό για μένα, δεδομένου ακριβώ του πλαισίου μέσα στο οποίο βρίσκεται την Ισία. Άλλε προτεραιότητε, τα είπαν κι άλλοι, είναι δικαιοσύνη, αστυνομία, μεταρρυθμίσει δηλαδή εκεί, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει έχοντα υπόψη μα μόνο την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτά που είπε και η Φιλεύθερη συνάδελφοι, την ελευθερία έκφραση, τελειώνω πρόεδρε. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι στην καρδιά των διαπραγματεύσεων που γίνονται στα πλαίσια πραγματική εταιρική σχέση. Να δίνουμε και να παίρνουμε και όχι μέσα σε ένα πλαίσιο όπου δεν λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της Τινησίας. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, όλοι μιλάτε μισό λεπτό παραπάνω. Είναι άδικο για τους υπόλοιπους συναδέρφους. Η κυρία Λοχμπίλερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε ε, και εξ ονόματος της, ε, των ε, Πρασίνων στο, στην Επιτροπή μας σήμερα εδώ, θα ήθελα να θέσω τρία ερωτήματα. Ε, καταρχήν, ε, είπατε ότι ε, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σταθερότητα στη Λιβύη και είναι θετικό το γεγονός ότι έχουν βρει προστασία και επιτρέπεται σε αυτούς να δουλεύουν ένα εκατομμύριο πολίτες της Λιβύης. Θα ήθελα να ρωτήσω, η δική σας χώρα λοιπόν λαμβάνει επαρκή διεθνή υποστήριξη ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την επιβάρυνση αυτή λόγω των προσφύγων, για παράδειγμα στον τομέα της υγείας ή της εκπαίδευσης. Δεύτερο ερώτημα, ε, σε ό,τι αφορά τον τομέα της ασφάλειας. Ε, προφανώς είπατε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ε, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και προφανώς το υποστηρίζουμε αυτό και η κοινωνία των πολιτών της Ισίας υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση. Ωστόσο, ακούσαμε πως και από τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ό,τι αφορά την προστασία ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι δεν θα πρέπει να είναι υπερβολική η προσέγγιση τη κυβέρνηση. Για παράδειγμα στο νέο νομοσχέδιο υπάρχει ε, και κάποιε κάποιες διατάξεις ό,τι αφορά την προσβολή των ενόπλων δυνάμεων. Εκεί προβλέπονται λοιπόν ιδιαίτερα υψηλές κυρώσεις και βέβαια είναι και έχει ασκηθεί κριτική σε αυτή την προσέγγιση την οποία συμμεριζόμαστε και εμεί, Δηλαδή αναφέρεται για παράδειγμα ότι ενδεχομένως να υπάρχει κίνδυνος ε, ε, της εθνικής ασφάλειας αλλά δεν ε, ορίζεται πώς ε, Αυτό ορίζεται ακριβώ στο νομοσχέδιο. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε από τη δική σα πλευρά. Θα υπάρξει κάποιο νομοσχέδιο στο μέλλον το οποίο θα προ... σέβεται πραγματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρίτο ερώτημα. σε ό,τι αφορά του μετανάστε προ στην Ευρώπη υπάρχουν υπάρχει μια συγκεκριμένη ε, ε, πολιτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακούσαμε πρόσφατα ότι ε, θέλει να δημιουργήσει κάποιες βάσεις στις αραβικές χώρες για drones, για μη επαντρωμένα δηλαδή αεροσκάφη. Ποια είναι η δική σας άποψη. κύριος Μποργέζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω κύριε Πρωθυπουργέ στο Κοινοβούλια, όμως, σας ακούσαμε με μεγάλη ικανοποίηση ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα καταπολεμήσετε την τρομοκρατία που είναι μία ε, μάστιγα που ε, ε, έπληξε τη χώρα σας ιδιαίτερα μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο Μουσείο του Μπαρντό. Θα θέλαμε να ε, συλληπιθούμε και τις οικογένειες των θυμάτων. Άρα η κυβέρνηση της Τινησίας έχει αναλάβει και ερευνητικό έργο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για αυτή την αντίσταση από, πλευρά πλευράς Ιταλικών αρχών για να στείλουν τον υπόδικο αυτό, τον ύποπτο για την τρομοκρατική αυτή δραστηριότητα, ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί στη χώρα σας. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας και οι πληροφορίες σας σε σχέση με την ε, τρομοκρατική διείσδυση μέσω διακινητών και μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο, γιατί αυτό το ακούμε πολύ συχνά και ακούμε διαφορετικές εκδοχές από τις κυβερνήσεις της Δύσης που ασχολούνται με τον έλεγχο. Μας λένε πολλές φορές ότι υπάρχουν διεισδύσεις, άλλες φορές όχι. Ίσως εσείς βρίσκεστε σε καλύτερη θέση να μας δώσετε ορισμένες ενδείξεις λόγω γειτονίας και ιδιαίτερα γειτονίας με τη Λιβύη. Ο Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα στη Επιτροπή, ενώπιον της Επιτροπής ΑΦΕΤ και των δύο υποεπιτροπών ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ασφάλειας. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας ε, στο, στο δραματικό θέμα της μετανάστευσης πώς μπορούμε να αποτρέψουμε κατά κάποιο τρόπο τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει υποδομή έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην θέλουν να μεταναστεύσουν. Όταν βρίσκονται στη Μεσόγειο δεν μπορούμε παρά να διασώσουμε τη ζωή τους, να σώσουμε ζωές. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα στην πηγή του. Πώς μπορείτε να προλαμβάνετε τέτοιες ε, ροές, γιατί όταν υπάρχουν πλέον τα μέσα που διαθέτουμε δεν είναι επαρκή. Επίσης η χώρα σας προβλέπει να ξεκινήσει συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διευκόλυνση του καθεστώτος των θεωρήσεων, γιατί υπάρχει μία συμφωνία και συμφωνία ενδεχόμενης επανεισδοχής, γιατί τα δύο αυτά ζητήματα συνδέονται. Θα ήθελα να ευχηθώ σε εσά και στη χώρα σας να μας δείξετε ότι υπάρχει μια ειρηνική μετάβαση προς τη δημοκρατία, ιδιαίτερα κατά αυτή την δύσκολη περίοδο για τη Βόρεια Αφρική, ιδιαίτερα μετά την ε, τρομοκρατική ενέργεια στο Μουσείο του Μαρντό. Ε, είχαμε θύματα και από τη δική μου εκλογική περιφέρεια. Ελπίζω να λύσετε αυτό το ζήτημα σύντομα. Κύριο Κάν. να σας καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ και χαιρετίζω και εγώ βέβαια την ε, βούληση που υπάρχει για να αναπτύξουμε στενότερες ε, σχέσει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και της χώρας σας και θα ήθελα να σα συγχαρώ βέβαια και την εκλογική διαδικασία και την δημοκρατική διαδικασία στη χώρα σα. Θα ήθελα να σα θέσω κάποια ευρύτερα ερωτήματα που αφορούν δηλαδή όλο το χρόνο τη Μεσογείου. Ε, πολλοί λοιπόν ανά τον κόσμο είχαμε ενθουσιαστεί με την Αραβική Άνοιξη και μετά είδαμε βέβαια να μετατρέπεται αυτή η Άνοιξη σε Αραβικό χειμώνα. Και ε, το, το ερώτημα εδώ είναι το, το πώς η δημοκρατία οδηγεί στην, ε, σε λιγότερη ασφάλεια δηλαδή το, ε, και το πώς τελικά ακούμε διάφορους να, να λένε ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ασφάλεια και όχι δημοκρατία. Πού μας οδηγεί λοιπόν μια τέτοια συλλογιστική. Από εκεί και μετά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν διάφορες χώρες σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του, ε, του εξτρεμισμού των ε, Ισλαμιστών. Ε, πού μπορεί κανείς λοιπόν να θέσει εδώ ένα όριο ανάμεσα σε τέτοιες πολιτικές της ασφάλειας και της καταπολέμησης της Και τέλος υπάρχει λειτουργούν, λειτουργεί το τάσος πόλος έλξης για πολλούς ε, ανθρώπους. Ε, ε, πώς λειτουργεί λοιπόν ως πόλος έλξης και πώς μπορούμε να δώσουμε κι εμείς από την πλευρά μας ένα εναλλακτικό μήνυμα. Πώς μπορείτε εσείς κύριε Πρωθυπουργέ να μας βοηθήσετε στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ, λέω ο Νομίζω θαύμα έγινε που κάποιος δεν υπέρευε το όριο. Κύριος Φίσας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, Θαυμάζω τη χώρα σας και είμαι φίλος της Τινησίας. Παρακολουθώ τις προσπάθειές σας προκειμένου να είσαστε μια χώρα στην πρώτη γραμμή μεταξύ των αραβικών χωρών στο δρόμο για τη δημοκρατία. Συμμετέχω στην Επιτροπή για το Διεθνές Εμπόριο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ρωτάω, είσαστε έτοιμος να υπογράψετε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τινησία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούζο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό και να του πω ότι στηρίζουμε τη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα του μέσα στα τόσο δύσκολα πλαίσια με την τρομοκρατία κτλ. Έχετε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στον αγώνα σας κατά της τρομοκρατίας. Θέλω λοιπόν τρεις ερωτήσεις να σας κάνω. Πρώτον, πώς βρίσκεται η αστυνομία, ποιες είναι οι ικανότητες της αστυνομίας για να προστατεύει και τη δημοκρατία μέσα στο δύσκολο πλαίσιο. Δεύτερον, Λιβύη στηρίζεται τις προσπάθειες του Βραντίνου Λεόνου, του ειδικού πεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί λύση σε περιφερειακό επίπεδο. Και η τρίτη μου ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σας για την δράση αυτή που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ενδεχομένω μέτρα ακόμα και στρατιωτικά για να αναχαιτιστεί η μετανάστευση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο και θα θέσω ένα-δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Σας ε, καλωσορίζουμε εδώ. Είναι πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε θετικά. Ήμασταν πριν από την ε, εκλογική διαδικασία στη χώρα σας ε, και πραγματικά είδαμε ότι ε, ε, γίνεται ένα διεθνώς σημαντικό κέντρο για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις από όλες τις αραβικές χώρες. Πραγματικά χαιρετίζουμε αυτή την σταθερότητα που κατάφερε να εδραιώσει η χώρα σας, αλλά υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ατζέντα για την ασφάλεια, καθώς θα μπορούσε πραγματικά με διάφορους τρόπους να υπονομεύσει τις, τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και ούτω καθεξής. Οπότε θα ήθελα ήθελα να σας ε, ζητήσω λοιπόν εδώ ε, να ε, τονίσετε την, την σημασία τέτοιων δικαιωμάτων τόσο στην Τινησία όσο και γενικότερα στον αραβικό χώρο και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό το επίπεδο τόσο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, προσωπείτε την, την Ισία. Εάν μία ε, ευρωπαϊκή χώρα έστελνε κάποια αεροσκά... Ε, αεροσκάφη τα οποία θα κατέστρεφαν ορισμένα πλοία τα οποία είναι προσαρμοσμένα σε ένα λιμάνι δικό σας. Θα υποστηρίσατε μια τέτοια ε, ομή παραβίαση ε, της κυριαρχίας της Τινησίας ή ε, ε, τι θα κάνετε, θα προβαίνατε σε κήρυξη πολέμου, θα περιμένατε την κάποια επίσημη συνόμη από αυτή τη χώρα, τι θα κάνατε από την πλευρά σας. Δεύτερο ερώτημα, δεν θα ήταν καλύτερο για την Τινησία. να είναι μια καλή χώρα στο πλαίσιο της γειτονίας, στο πλαίσιο της Κυριναϊκής ή θα έπρεπε να θέσει περισσότερη έμφαση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο ε, Μπροκ, δεν μπορεί κανεί ε, να επιλέγει τι γειτονικέ του χώρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Κυρίε και κύριοι, θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη χώρα μου, την Τινησία. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και πριν να αρχίσω πείτε μου πόσο χρόνο έχω παρακαλώ. Όσο θέλετε, απαντά ο κύριος Μπρόκ. Ωραία, να, διάκριση. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι η κατάσταση στην ε, την Ισία αυτήν τη μεταβατική περίοδο είναι πολύ ιδιαίτερη. Καταφέραμε να πετύχουμε την ε, μεταπολίτευση. Ήταν δύσκολο Τρία χρόνια και κάτι μήνες μας πήρε για να ολοκληρωθεί αυτή η αλλαγή, η οποία έγινε κάτω από καλές συνθήκες, όπως είπατε κι εσείς. Δεν ήταν τέλεια, αλλά καταφέραμε η μετάβαση αυτή να γίνει κάτω από τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες και είμαστε ικανοποιημένοι που πετύχαμε αυτό το στάδιο πολιτικής μετάβασης. Πολύ σημαντικό για την ιστορία της χώρας μας. Είναι η πρώτη φορά που η μετάβαση αυτή γίνεται κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η δουλειά όμως μόλις άρχισε. Μένουν πολλά να γίνουν ακόμα, σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια μεγάλη πολιτική πρόκληση. Γιατί έχουμε ένα σύνταγμα, βεβαίως. Αλλά το να θέσουμε σε εφαρμογή το περιεχόμενο αυτού του συντάγματος αποτελεί για μας μια μεγάλη πρόκληση, γιατί έχει δυσκολίες και κινδύνους. Στα πλαίσια λοιπόν της δράσης της κυβέρνησης αυτής της δεύτερης δημοκρατίας προσπαθούμε να τηρήσουμε απόλυτα το περιεχόμενο του συντάγματος αυτού. Ένα περιεχόμενο το οποίο διασφαλίζει δικαιώματα και ελευθερίες για τους την ίσιους, όπως συμβαίνει σε κάθε δημοκρατική χώρα. Και εδώ ακριβώ είναι που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο του συντάγματος αυτού. Έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μένουν όμως πολλά να γίνουν. Όλα όσα προβλέπονται στο σύνταγμά μας πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή. Δικαιοσύνη, ε, συνταγματικό συμβούλιο, συμβούλιο επικρατείας δηλαδή, και όλοι αυτοί οι δημοκρατικοί θεσμοί που προβλέπονται στο Σύνταγμα μένει να λειτουργήσουν σύμφωνα με το Σύνταγμα. Έχουμε ήδη προετοιμάσει τη βάση προκειμένου να μπούμε σε αυτήν την ε, μακρά διαδικασία και σε βάθος αλλαγή. Πολιτικά μιλώντας λοιπόν έχουν ανοίξει πολλά εργοτάξια για να το πω έτσι και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράμε και σε συνεργασία και με όλες τις άλλες φίλες χώρες που μας στηρίζουν στη μεταβατική αυτή περίοδο. Το εργοτάξιο της ασφάλειας είναι πάρα πολύ λεπτό και πάρα πολύ σημαντικό. Όπως το γνωρίζετε, δεν μπορούμε να μιλάμε για ελευθερίες και δημοκρατία αν δεν έχουμε ασφάλεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και για επενδύσεις χωρίς ασφάλεια. Συνεπώς, η πρώτη μας επιλογή, μία από τις πρώτες επιλογές που έκανε η κυβέρνηση αυτή, είναι η ασφάλεια ακριβώς. Και εργαζόμαστε εκπονούμε στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κάτι το οποίο είναι για μας προτεραιότητα. Όπως διαπιστώσατε και όπως το είπαν και ορισμένοι, η τρομοκρατική ενέργεια εκείνη, η επίθεση τρομοκρατική η οποία έλαβε χώρα στον Παρντό, είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι οι τρομοκράτες, εκείνοι που δεν θέλουν το καλό της την και προέβησαν στην επιθετική αυτή πράξη, μα ζηλεύουν σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε. Ζηλεύουν την Τινησία η οποία καταφέρνει να κάνει τόσο σημαντικά βήματα προς τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Η επίθεση αυτή, η βάρβαρη, στο μουσείο ήταν για να χτυπήσει όσο γίνεται περισσότερες εθνικότητες. Αυτός ήταν ο κακός στόχος, να πλήξουν την Τινησία στον τομέα εκείνο που είναι προτεραιότητα, που αποτελεί κινητήριο δύναμη της οικονομίας της. Θέλησαν να χτυπήσουν όσο γίνεται περισσότερες υπηκότητες, ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο γίνεται πιο εντυπωσιακά. Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι έχουμε τέτοιες συμπεριφορές, γι' αυτό έχουμε εκπονήσει στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να επιτεθούμε εμείς στην τρομοκρατία. Και έχουμε δύο δράσεις για να ε, για να διαλύσουμε. Πρώτα απ' όλα διαλύσαμε μια πολύ σημαντική οργάνωση. Ο αρχηγός της κατάφερε να ξεφύγει όμως διαλύσαμε την οργάνωση αυτή. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του αγώνα μας. Ο στρατός επίσης επιτέθηκε σε μια ομάδα εκεί που είχε την έδρα της. Κάτι πολύ καλό για το ηθικό. Τώρα οι τρομοκράτες γνωρίζουν ότι δεν είναι αυτοί που μπορούν να προχωρήσουν σε επιθετικές ε, πράξεις. Η αστυνομία και ο στρατός μπορεί να τους επιτεθεί και να τους ε, αδρανοποιήσει. Αυτά που κάναμε λοιπόν το τελευταίο καιρό αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την αποσταθεροποίηση των τρομοκρατών. Στο οικονομικό επίπεδο τώρα. Εδώ προετοιμάζουμε ένα σημείωμα προσανατολισμού για την προετοιμασία της νέας μας στρατηγικής που θα αρχίσει το 2016 και πάει μέχρι το 2020. Πρόκειται για ένα πενταετές ε, πρόγραμμα όπου αναφέρονται κύριες επιλογές και οι κύριοι άξονες της χώρας για την επόμενη αυτή περίοδο. Βάσει λοιπόν αυτού του σημειώματος προσανατολισμού που θα συζητηθεί σε όλα τα επίπεδα, προβλέπεται μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία θα αποτελείται από δύο άξονες. Αναπτυξιακό πρόγραμμα πρώτα απ' όλα, όπου έχουμε επιμέρους προγράμματα υπέρ των περιφερειών και όπως γνωρίζετε έχουμε εντοπίσει 14 περιφέρειες στη χώρα που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Προβλέπεται και από το Σύνταγμα να ευνοηθούν οι περιφέρειες αυτές σε σχέση με άλλες προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά που έχουν απέναντι σε άλλες περιφέρειες. Καθυστέρηση η οποία συσσωρεύτηκε τα τελευταία χρόνια. Για κάθε περιφέρεια λοιπόν θα υπάρχει περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τις ικανότητες που έχει η κάθε περιφέρεια. Επιπλέον από τα περιφερειακά αυτά ειδικά προγράμματα για να δοθεί η όθηση στην ανάπτυξη των λιγότερο ευνομένων περιοχών, υπάρχουν και καμιά δεκαπενταριά διαρθρωτικά προγράμματα, τα οποία θα καλύψουν το σύνολο της εθνικής επικράτειας. Προβλέπεται στο τέλος της προετοιμασίας μέχρι τα τέλη του 2015 να οργανώσουμε και μια διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών και των αναπτυξιακών αυτών περιφερειακών προγραμμάτων. Το άλλο όμως, ο άλλος άξονας, πιο σημαντικός που εκ θα λάβει η χώρα με τα αναπτυξιακά προγράμματα είναι οι μεταρρυθμίσεις μας. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη αρχίσει. Τράπεζες, φορολογία, επενδυτικός κώδικας, κοινωνική ασφάλιση, όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν πολύ σημαντικές δράσεις οι οποίες πρέπει να λάβουν χώρα εκ παραλλήλου με τα αναπτυξιακά προγράμματα. Αυτά προετοιμάζουμε λοιπόν στον οικονομικό τομέα. Και τώρα θέλω να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις που τέθηκαν από τους ευρωβουλευτές. Το πρόβλημα της μετανάστευσης. Πολλοί από σας αναφερθήκατε σε αυτό. Η Ισία το Φεβρουάριο του 2011 έζησε μια κατάσταση παρόμοια με την σημερινή. Θυμόσαστε ότι σε δύο μέρες πάνω από 20.000 Τινήσοι έφυγαν και πήγαν στην Ιταλία. Ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την Ιταλική κυβέρνηση τότε. Τότε λοιπόν διαπραγματευτήκαμε και προχωρήσαμε σε συμφωνία με την Ιταλική κυβέρνηση που ισχύει ακόμα και σήμερα. Πρόκειται για τον εντοπισμό των ανθρώπων που βρίσκονται επί τόπου και να έχουμε σχέσεις στα πλαίσια των συμφωνιών και να επαναπατριστούν όσοι είναι την ίση. Η συμφωνία αυτή ισχύει ακόμη και σήμερα. Τα τελευταία νούμερα που μου δόθηκαν λένε ότι το 2014 από τους 1.200 ίσιους που προσπάθησαν να μεταναστεύσουν στην Ιταλία, 1.100-1.150 επαναπατρίστηκαν, επέστρεψαν και τους ανέλαβε η, την Ισιακή κυβέρνηση, η οποία επαλήθευσε περί πρόκειται και τους ένταξε και πάλι στην ε, κοινωνία και στη χώρα. Θέλω να απαντήσω και σε μια ερώτηση που έθεσαν διάφοροι ευρωβουλευτές που ρώτησαν τι μπορούμε να κάνουμε για να εμποδίσουμε αυτήν την ροή, τη μεταναστευτική και τι μπορούμε να κάνουμε για να ενσωματώσουμε και πάλι στη χώρα αυτούς που επαναπατρίζονται. Γιατί αν δεν έχουμε λύση για να τους επαναπατρίσουμε, για να τους εντάξουμε και πάλι στη χώρα... Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να εμποδίσουμε τη μετανάστευση είναι να βρούμε λύσεις επιτόπου. Να δημιουργούμε δηλαδή προγράμματα, ε, τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες βοηθούν τον κόσμο να βρει δουλειά στη χώρα του να έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποια προοπτική στη χώρα τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Και στη συνέχεια πρέπει από τη στιγμή που γίνεται η μετανάστευση, απαξί και υπάρχει επαναπατρισμός, αυτό που κάναμε και εμείς δηλαδή με την Ιταλική κυβέρνηση, συμφωνία, στη συνέχεια να δίνουμε δυνατότητες στους ανθρώπους αυτούς να έχουν ευκαιρίες πίσω στη χώρα τους. Και έχουμε προγράμματα τα οποία είναι πετυχημένα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που επαναπατρίστηκαν, αλλά μετά έφυγαν. Έχουμε μερικέ τέτοιε περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται, ξαναφεύγουν. Θέλουμε λοιπόν να προετοιμάζουμε τέτοια αναπτυξιακά προγράμματα, σαν και αυτά που σας είπα για τις 14 περιφέρειες, ακριβώς ώστε οι πολίτες να έχουν ενδιαφέρον να μείνουν, να έχουν λόγο να μείνουν στη χώρα τους και να μην θέλουν να φύγουν. Στο άγνωστο. Το κίνδυνος της τρομοκρατίας μέσω της μετανάστευσης, ναι, μπορεί να υπάρχει. Ο τρομοκράτης που συνελήφθη στην Ιταλία και που συμμετείχε στην επίθεση στον Παρδό, είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν στην Τινησία και έφυγε προς τη Λιβύη. Προχτές συλλάβαμε και τον τέταρτο τρομοκράτη, ο οποίος αναμίχθηκε επευθεία στην επίθεση αυτή. Στη Λιβύη κι αυτός. Ο κίνδυνος λοιπόν να ανακατευτούν οι τρομοκράτες με τα πλήθη που φεύγουν να μεταναστεύσουν ε, υπάρχει. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να φροντίσουμε οι τρομοκράτες και οι μετανάστες να παραμένουν στη χώρα τους. Κάτι άλλο τώρα που με ρώτησαν πολύ για τη θέση της Τινησίας όσον αφορά την δράση που σκέφτεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει τα κύματα αυτά, τα διαδοχικά κύματα μεταναστών. Η θέση της Τινησίας ήταν πάντα η ίδια. Το κάναμε και με την Ιταλία. Παρέμβαση στρατιωτική για να λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί με αναπτυξιακές δράσεις ή με προληπτικές δράσεις είναι τρέλα. Κάθε στρατιωτική παρέμβαση μας βρίσκει αντίθετους. Είμαστε κατά κάθε στρατιωτικής δράσης, είτε για να λυθεί ένα πολιτικό ζήτημα, είτε για να λυθεί το μεταναστευτικό της λαθροδιακίνησης. Ρωτήσατε και κάτι για τη θέση της Τινησίας όσον αφορά την Λιβική σύγκρουση. Η κατάσταση για μας είναι σαφής στη Λιβύη. Είμαστε κατά κάθε στρατιωτική παρέμβαση για να λυθεί το Λιβικό. Η σύγκρουση εκεί είναι πολιτική και δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο μέσω πολιτικής λύσης, μέσω διαπραγματεύσεων. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Η προσέγγιση της Τινησίας με τη Λιβύη δεν είναι αλήθεια. Κάθε αυτή που κάναμε όλο αυτό τον τελευταίο καιρό, συναντηθήκαμε και με την κυβέρνηση της Τρίπολης και του Δουμπρούκ. Και προσπαθήσαμε στα πλαίσια την Ισιακής πρωτοβουλίας σε άμεση συνεργασία βέβαια με τα Ηνωμένα Άθνη, προσπαθήσαμε να υπάρξει μια προσέγγιση ανάμεσα στις θέσεις των δύο πλευρών, των δύο κυβερνήσεων. Και για μας είναι σημαντικό η λύση της Λιβύης, η λύση του Λιβικού να έρθει γρήγορα, με πολιτικό τρόπο και με διαπραγματεύσεις. Με υπομονή πιστεύω ότι μπορούμε να λύσουμε τη σύγκρουση αυτή. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω μια που εντάξει, χρόνο δεν μπορεί να έχω και περιόριστο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για το ενδιαφέρον που δείχνουν απέναντι στην Τινησία. Η Τινησία είναι μια νέα δημοκρατία. Πολλά μένει να γίνουν ακόμα σε όλα τα επίπεδα, στο πολιτικό, στο οικονομικό, στο κοινωνικό, στο επίπεδο της ασφάλειας. Βασιζόμαστε πάρα πολύ στη συνεργασία μαζί σας και στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους ιδιαίτερους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να μας βοηθήσετε να πετύχουμε στην μετάβασή μας αυτή, προκειμένου την Ισία να είναι ένα παράδειγμα να δείξουμε και στους άλλους ότι πολιτικά μπορούμε να πετύχουμε σημαντικές αλλαγές χωρίς να χρειάζονται άλλα μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ ε, θερμά. Νομίζω πως ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντησή μας. Ε, Εύχομαι να περάσετε όμορφα στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.